υπάρχουν και, μετα... και οδηγοί από τρίτες χώρες που προφανώς ε, θα βρεθούν σε καλύτερη ε, μοίρα σε σχέση με τους κοινοτικούς οι οποίοι θα ήταν πολύ πιο θα έπρεπε να ε, εφαρμόσουν κανόνες πολύ πιο αυστηρούς. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, ναι. το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα το πρωί είναι μια έκθεση της κυρίας Ρενάτε Ζόμερ για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Τον λόγο τον έχει η συγγήτρια, η κυρία Ζόμερ. Περιμένω να ησυχάσει λίγο η αίθουσα. Θα δώσω όμως αμέσως το λόγο στην κυρία Ζόμερ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τέσσερα λεπτά και άλλα δύο λεπτά. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν έξι λεπτά γιατί το θέμα αυτό είναι τόσο περίπλοκο που πιστεύω ότι θα μας χρειαστεί αυτός ο χρόνος. Το σημαντικό λοιπόν αυτό θέμα αφορά τα τρόφιμα και την απόφαση του καταναλωτή να τα αγοράσει βάσει σωστής ενημέρωσης. Μιλάμε λοιπόν για την επισήμανση και τις ετικέτες. Όσον αφορά τους εμπόρους και όσον αφορά τους καταναλωτές, υπάρχει πληθώρα νόμων, ρυθμίσεων οι οποίες ε, είναι σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό πολλές φορές μας οδηγεί σε ένα περίπλοκο σύστημα που έχει σαν συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού της ευρωπαϊκής αγοράς. Προσπαθούμε λοιπόν να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση με καλύτερη ενημέρωση, με εναρμόνιση, με μείωση της γραφειοκρατίας και με καλύτερες και πιο σαφείς ε, νομοθετικές ρυθμίσεις. Ο καταναλωτής σήμερα θέλει να έχει καλύτερη ενημέρωση και να μπορεί, παραδείγματο χάρη, να έχει ευανάγνωστες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι ε, γραμμένες με μικρά γράμματα, τόσο μικρά που κανείς δεν μπορεί να τα διαβάσει. Το 80% των τροφίμων θα πρέπει να καλυφθούν από αυτές τις ρυθμίσεις γιατί σήμερα βλέπουμε ότι η ισχύουσα κατάσταση είναι αντίθετη με την προσπάθειά μας να εναρμονίσουμε την ενιαία αγορά και να δώσουμε σωστή, κατανάλωση, σωστή ενημέρωση στους καταναλωτές. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ορίσουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ε, ε, πληροφορίες οι οποίες να είναι σαφείς, να είναι ευανάγνωστες, να μπορεί κανείς να τις διαβάσει χωρίς να πρέπει να κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια όσον αφορά παραδείγματο χάρη τις ποσότητες, να μην υπάρχουν μόνο ποσοστά αλλά να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ενδείξεις του βάρους σε χιλιόγραμμα παραδείγματο χάρη. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι κατανοητές. Αυτό το κιλο τζάουλ το οποίο κανείς δεν καταλαβαίνει να σταματήσει να είναι εγγεγραμμένο σε όλες τις ε, ετικέτες αλλά να μιλάμε για θερμίδες. Οι θερμίδες οι οποίες πραγματικά είναι κατανοητές σε όλους και όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να αναγράφονται με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε τις ε, καταχρήσεις, τις εσφαλμένες ας πούμε πληροφορίες για προϊόντα που είναι απομιμήσεις άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούν παραδείγματος χάρη κάποιες πρωτεΐνες που δεν είναι όμω οι πρωτενε του κρέατος το οποίο θέλει να αγοράσει ο καταναλωτή ή που είναι ένα υποκατάστατο κρέατο ή υποκατάστατο τυριού. Επαναλαμβάνω, ε, οι ενδείξει θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες. Μιλάμε παραδείγματος χάρη για στοιχεία που να μπορούν να είναι κατανοητά και τα ίδια πάντα, όπως θερμίδες ανά χίλια γραμμάρια, παραδείγματος χάρη, ή 100 γραμμάρια, συγκεκριμένες ενδείξεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν τα ανώτατα όρια για τα λύπη ή για άλλα συστατικά τα οποία θέλουν να γνωρίζουν οι καταναλωτές. Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να υπάρχουν ακριβή στοιχεία και όχι η επιπλέον επιβάρυνση των διαδικασιών. Σκοπός μας δεν είναι να κατατάξουμε τα τρόφιμα σε καλά ή κακά τρόφιμα, αλλά να μπορεί κάποιος να γνωρίζει τι ακριβώς περιέχει ένα προϊόν το οποίο αγοράζει. Το θρεπτικό προφίλ, τις θρεπτικές ουσίες, τα συστατικά, τις πρόσθετες ουσίες και ε, που δεν είναι λόγο, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο κατηγορίες ειδών διατροφής, τα καλά και τα κακά, τα χρήσιμα και τα μη χρήσιμα. Που δεν λόγο, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες διακρίσεις, όλα τα προϊόντα, ακόμα και αυτά τα οποία περιέχουν ε, κάποιες ουσίες που σήμερα είναι λιγότερο αν θέλετε καλές από διατροφική άποψη θα πρέπει να μπορούν να αναγράφονται. Οι χρωστικές ουσίες, τα αρώματα, η ζάχαρη. Σήμερα βλέπουμε ότι οι θρεπτικές ουσίες δεν περιγράφονται με σωστό τρόπο. Παίρνετε μια κατηγορία καταναλωτών, όπως παραδείγματο χάνει οι γυναίκες 40 ετών και οι θρεπτικές αναλογίες και ποσοστά απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε αυτή την κατηγορία. Κάτι το οποίο είναι λανθασμένο. Δεν είναι ίδιε οι θρεπτικέ ανάγκε και οι διατροφικέ ανάγκε όλων των κατηγοριών. Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε όλε αυτέ τι κατηγορίε. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε και κάποιε κατηγορίε εξαιρέσεων για τρόφιμα τα οποία σήμερα δεν καλύπτονται από καμία νομοθεσία. Οι παραγωγοί, οι κατασκευαστές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους λοιπόν όλες αυτές τις νέες ρυθμίσεις και το ερώτημα είναι αν ο καταναλωτής θέλει παραδείγματο χάρη να γνωρίζει την προέλευση όλων των ε, θρεπτικών ε, ε, αυτών συστατικών, όλων των προϊόντων που αγοράζει. Θα πρέπει βεβαίως πολύ σύντομα να γίνει και μία μελέτη αντικτύπου και συνεπιών και να προσαρμόσουμε κατόπιν ε, την κατάσταση βάση αυτής της μελέτης αντικτύπου. Τελειώνω κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Δεν είναι σκοπός ε, κανενός νομοθέτη να αποφασίσει στη θέση του καταναλωτή, στη θέση του Ευρωπαίου πολίτη. Σκοπός μας όμως και καθήκον μας είναι να ενημερώσουμε και να δίνουμε ακριβείς, κατανοητές και ευανάγνωστες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ, διακόπτη Πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Ο κύριος Ντάλι έχει το λόγο. Thank you very much, President. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι αγοράζουν και τι τρώνε. Με τον τρόπο αυτό είναι πιο εύκολο για αυτούς να επιλέξουν την δίαιτά τους και για τους εαυτούς τους και για την οικογένειά τους ανάλογα με τις ανάγκες τους, με τις επιθυμίες τους και με τους στόχους τους. Οι πολίτες, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα για σωστή πληροφόρηση. Θα ήθελα να απευθύνω μία κλίση και στους βουλευτές να έχουν αυτό στο μυαλό τους καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Τώρα, Επί της ουσίας θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία, την κυρία Σόμερ, διότι συνέταξε την έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους κοιόδης εισηγητές. Ε, αντιμετωπίζω με κατανόηση τα σχόλια όλων, όχι όμως ε, δεν μπορώ να πω ότι δέχομαι και τις απόψεις τους. Θα ήθελα να τονίσω τα πιο βασικά θέματα τα οποία καλύπτει η πρόταση και οι προτινόμενες τροπολογίες. Το θέμα της υποχρεωτικής ε, συμπερίληψης κάποιων προφοριών στην δικαιοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, υπάρχει μια ε, αίτηση, ένα αίτημα να συμπεριλαμβάνονται κάποιες υποχρεωτικές πληροφορίες για κάποια τρόφιμα. Η Κομισιόν μπορεί να δεχτεί εν μέρη την τροπολογία όσον αφορά την προέλευση της πληροφορίας για την προέλευση ε, οι πληροφορίες που αφορούν ένα, ένα και μόνο ένα προϊόν το οποίο αποτελείται από ένα και μόνο υλικό, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δεχτούμε. Οποιαδήποτε υποχρεωτική ε, αναγραφή για, την, για την προέλευση θα πρέπει να εξεταστεί ε, ξεχωριστά. Κάθε αίτημα και κάθε προϊόν ξεχωριστά. Εμείς ε, θεωρούμε ότι οι καταναλωτές ε, είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν συζητάμε η προστασία των καταναλωτών. Ε, και θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουμε μετρήσιμα αν θέλετε, κριτήρια για την εφαρμογή της, των κανόνων. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με τους βουλευτές όσον αφορά τα προϊόντα απομίμησης. Θα πρέπει να ε, απαγορεύσουμε τέτοιου είδους πρακτικές. Όμως η εισαγωγή ενός ορισμού ε, για τα προϊόντα αυτά θα, θα δημιουργούσε νομικά προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, βρούμε κάποιες, ε, κάποιες ενδείξεις οι οποίες να δίνουν σαφείς ε, πληροφορίες στους καταναλωτές. Επίσης, συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικές αναγραφές όσον αφορά την διατροφική αξία των προϊόντων και όχι μόνο στα προς προσυσκευασμένα αλλά και στα άλλα προϊόντα τα οποία αγοράζουν καπευθείαν. Επομένως δεν συμφωνούμε με τις ε, τροπολογίες που περιορίζουν το ε, πεδίο εφαρμογής ε, της, του κειμένου. θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε ένα σύστημα που να έχει κάποιες συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες και από εκεί και πάρει τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν περαιτέρω διατάξεις. Επίσης, στο θέμα των για τα διατροφικά προϊόντα, ε, ήθελα να πω ότι συνειδητοποιούμε απόλυτα ότι κάποια από αυτά τα οποία αναφέρα, γράφονται πάνω στη συσκευασία είναι παραπλανητικά. Γιατί ε, ε, κάποια είναι εν μέρη ε, αληθή και κάποια κρύβουν κάποια πράγματα από τους καταναλωτές. Ε, διάφορες ε, δηλώσεις ε, γίνονται εξ ονόματος του κατασκευαστή για να πουλήσει περισσότερα προϊόντα. Εμείς δεν επιβάλλουμε το διατροφικό προφίλ των προϊόντων. Το διατροφικό προφίλ το προωθούν οι κατασκευαστές για να έχουν οι καταναλωτές κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες. Η εμφάνιση του διατροφικού προφίλ δεν περιορίζει, αν θέλετε, την αξία των των προϊόντων. Οι κατασκευαστές προϊόντων μπορούν να παράγουν και να συσκευάζουν με τον τρόπο τον οποίο, όχι να παράγουν, να συσκευάζουν με τον τρόπο τον οποίο θέλουν. Όμως είναι άδικο για τους ε, καταναλωτές να διαβάζουν ε, δηλώσεις που μπορούν να τους παραπλονίσουν. Είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε έντιμες ε, και σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές για τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουν. Ο κανονισμός για τις δηλώσεις αυτές, αν θέλετε, έχει υιοθετηθεί μετά από συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της κοινότητας και η νομοθεσία αυτή παραμένει ενισχύ. Βέβαια, τα διατροφικά προφίλ θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε με ένα ανοιχτό μυαλό και ε, θα εξετάσουμε θετικά κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν παραδοσιακά προϊόντα και που παίζουν ένα σημαντικό διατροφικό ρόλο. Με βάση όλα αυτά θα ήθελα να σας, ε, να σας ζητήσω να υποστηρίξετε την πρόταση της Κομισιόν για να ε, έχουμε μια σωστή βάση για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας ε, και προσβλέπω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Κυρία Σαλδεμόζου, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή ΙΜΚΟ έχει προετοιμάσει μια έκθεση και μια γνωμοδότηση για την πρόταση κυρία Σόμερ. Θεωρούμε ότι πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει την ε, προσπάθεια αυτή έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να κάνει εν γνώση του την ορθή επιλογή. Συμφωνούμε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν σαφή μηνύματα, κατανοητά μηνύματα και ότι η εσωτερική αγορά θα πρέπει να λειτουργήσει με κοινού κανόνες. Συμφωνούμε λοιπόν απολύτως όσον αφορά την εφαρμογή, την πρακτική εφαρμογή αυτών των προτάσεων. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ αλλά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος συμφώνησε με τις προτάσεις αυτές. Ζητούμε από την εισηγήτρια να μην αγνοήσει το γεγονός ότι εδώ πρόκειται για ένα εργαλείο για τους καταναλωτές και όχι για τους ε, κατασκευαστές. Εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας... Ο κύριος Ταραμπέλα. Είμαι θυμωμένος, διότι θέλω να περιοριστώ στην 101 για τη χώρα προέλευσης. Εμείς είχαμε ζητήσει μια, διαχωρισ... χωρισμένη ψηφοφορία. Με δύο λόγια, χώρα προέλευσης είναι η χώρα τελευταίας μεταποίησης και όχι η χώρα αρχικής προέλευσης. Από εκεί που έρχονται τα λαχανικά, για παράδειγμα, πρώτες ύλες το Κοινοβούλιο αρνήθηκε αυτή μας την ε, πρόταση, χωρίς όμως να μου αναφερθεί, να στηρίξει την αποφασίση σε ένα συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού. Ε, μου είπαν ότι βασιζόμαστε στο, στα ήθη, στο έθιμο του Κοινοβουλίου μάλλον. Όμως, αυτό θα επηρεάσει την τελική απόφαση που θα βάλει το Κοινοβουλίο. Συνεπώ, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ να ζητήσετε από τι υπηρεσίε σα να διορθωθεί το θέμα μέσα στι επόμενε 24 ώρε να ξαναδούν οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου αυτή την πρόταση και το, τα επιχειρηματά του. Ευχαριστώ πολύ. Εξ των πολιτικών ομάδων, ο πρώτο ομιλητή για το ΕΛΚ είναι ο κύριο Λίζε. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ζόμερ για την σκληρή της εργασία, την εργασία αυτή η οποία τελικά οδήγησε σε κάποιες αβάσιμες ε, κριτικές. Σε πολλά από αυτά τα θέματα συμφωνούμε τελικά, γιατί όλοι θέλουμε να υπάρχει καλύτερη επισήμανση των ε, τροφίμων. Ένα τυρί θα πρέπει να έχει σαν κύριο συστατικό το γάλα. Αν υπάρχουν άλλες ουσίες που δημιουργούν πρωτενε μέσα στο τυρί, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται με πάρα πολύ κατανοητό τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που όλοι το θέλουμε. Επίσης όλοι θέλουμε με ενιαίο τρόπο να πληροφορήσουμε τον καταναλωτή. Στη Γερμανία, αλλά πιστεύω και σε άλλες χώρες, υπάρχουν κάποιες Πληροφορίε οι οποίε δεν είναι κατανοητές. Παραδείγματο χάρη, μιλάμε για τις θερμίδες την ίδια ώρα. Όταν μιλάμε για τις θερμίδες βλέπουμε να αναγράφονται kilojoule. Τα kilojoule καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κατανοητά και δεν μπορεί κανένας καταναλωτής να καταλάβει σε τι αναφέρεται. Θα πρέπει λοιπόν και για αυτό το θέμα αλλά και για άλλα οι πληροφορίες να δίνονται με έναν ευανάγνωστο και ενιαίο τρόπο. Επίσης η συζήτηση που οδήγησε πολλές αντιπαραθέσεις αφορά και κάποιες εθνικές ευαισθησίες όπως το τυρί για τους Γάλλους, τα αρτοσκευάσματα για κάποιες άλλες χώρες. Ζητώ λοιπόν να στηρίξετε τις τροπολογίες του ΕΛΚ στον τομέα αυτό των κάποιων παραδοσιακών προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυρία Βόλμαρτ έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ε, είναι πολύ επίμαχη αυτή η πρόταση και πολύ περιπλοκή. Ω σκιώδη ηγητρία τη ομάδα μου, θα ήθελα να πω ότι η βασική μου αρχή είναι να ρωτήσουμε τον εαυτό μα ποιε πληροφορίε χρειάζονται οι καταναλωτέ και πώ εμεί μπορούμε να του παρέχουμε τον καλύτερο τρόπο. Αυτή τη ε, στιγμή ε, τρώμε πάρα πολλά λίπη, πολύ αλάτι και πολύ ζάχαρη. Αυτό οδηγεί σε διαβήτη, ε, καρδιακά προβλήματα, καρκίνους, ε, ασθένειες του ύπατος κλπ. Θα πρέπει λοιπόν οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζουν καλά το, τη διατροφική αξία αυτών που τρώνε. Βέβαια αυτό δεν είναι πανάκια, αλλά θα τους βοηθήσει να συγκρίνουν προϊόντα και να έχουν μια συνολική άποψη αμέσως. Θα μπορέσουν δηλαδή να έχουν καλύτερο έλεγχο αυτού που τρώνε. Προτείνω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα χρωματικών κωδικών για να ενημερώσουμε τους καταναλωτές αν το προϊόν που αγοράζουν είναι, έχει ψηλή, μέση ή χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι κλπ. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ε, ιδιαίτερα μεταπημένα προϊόντα, ε, έτοιμες τροφές, έτοιμα τρόφιμα κλπ. Ε, γιατί πολύ συχνά οι καταναλωτές μας δεν γνωρίζουν ή παραπλανούνται αυτό δεν θα εφαρμοζόταν στο γερμανικό ψωμί, δεν θα εφαρμοζόταν ούτε στο τυρί, ούτε στο ε, αλκοόλ, ούτε στους χυμούς μήλου. Ε, το έχω πει αυτό και έστειλα και ένα mail. Σας διαβάστε το πριν αποφασίσετε για να ξέρετε τι προτείνουμε. Μην ακούτε παραπλανητικές φωνές του, των λόμπις των, ε, των επιχείρησεων του κλάδου. Επίσης ζητήσαμε ε, υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής διότι οι κατανοητές θέλουν να ξέρουν πού έρχονται, όλο και περισσότερο θέλουν να ξέρουν πού προέρχονται τα τρόφιμά τους. Αυτό βέβαια δεν θα είναι πάντοτε ε, δυνατό, αλλά για απλά προϊόντα, μοναδία προϊόντα, θα έπρεπε να γνωρίζουν οι κατανοητές από πού προέρχονται γιατί είναι πρώτες ύλες. Αυτό ήδη γίνεται και στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και στο ψάρι. Εκεί είναι δυνατόν να γίνει. Τώρα βέβαια σε μεταποιημένα και σύνθετα προϊόντα είναι πιο περίπλοκο. Γι' αυτό το λόγο εμείς το προτείνουμε μόνο για τα ψάρια, τα κρέατα και τα πουλερικά σε με, μεταποιημένα τρόφιμα. Ε, ε, εν γέννη, ε, οι κανόνες αυτοί έχουν σχέση με τι επιλογέ των καταναλωτών. Ας είμαστε σοβαροί για μία φορά. οι πράξεις ακούγονται περισσότερο από τα λόγια. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Καπράντη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο για όλες αυτές τις ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ και την κυρία Σόμερ για τα όσα έκανε σαν εισηγήτρια. Έχω την εντύπωση μετά από ένα χρόνο που είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου, ότι η ιδέα ότι μπορούμε να επηρεάσουμε με μια απλή νομοθεσία τη συμπεριφορά εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών είναι μια ιδέα που με ενθουσιάζει. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η συμπεριφορά των πολιτών και μιλάμε για 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Οι διατάξεις όσον αφορά λοιπόν την επισήμανση πιστεύω εγώ ότι θα έχουν περιορισμένες συνέπειες. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές την ίδια ώρα. Συμφωνώ απολύτως ότι ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες βάσιμες, σωστές. Και προς το παρόν βλέπουμε ότι στη δεύτερη ανάγνωση αν το κείμενο αυτό περάσει ως έχει, ο καταναλωτής στην Ευρώπη θα έχει περισσότερες πληροφορίες και πιο ορθές. Την ίδια ώρα όμως θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες και στον τομέα της ε, ενημέρωσης, της γενικότερης και της εκπαίδευσης των Ευρωπαίων πολιτών. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καθοριστικός. Μπορούμε εμείς να πιέσουμε, να υποχρεώσουμε τους ε, Ευρωπαίους να κάνουν υγιείς επιλογές. Είμαστε φιλελεύθεροι και θεωρούμε ότι ο Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να επιλέξει εν γνώση του τι θέλει να αγοράσει. Και θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση γιατί πληθώρα πληροφοριών πολλές φορές είναι καταστροφική. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια μέση λύση μεταξύ των ε, εσφαλμένων ή ελλειπών πληροφοριών και του κατακλυσμού απληροφορίας. Ευχαριστώ πολύ για τους πράσινους, ο κύριος Κάλς Λίτερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η δύναμη του καταναλωτή στηρίζεται στις πληροφορίες που λαμβάνει. Εάν οι επιχειρήσεις δεν τους δίνουν τις κατάλληλες πληροφορίες, τότε όλη η εσωτερική αγορά θα καταρρεύσει, διότι οι καταναλωτές δεν θα έχουν εξουσία, δεν θα έχουν δύναμη. Οι, εξου... οι καταναλωτές έχουν κάποιες απαιτήσεις και θα πρέπει να ικανοποιήσουμε στον δυνατόν περισσότερες απαιτήσει των καταναλωτών. Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε τους καταναλωτές ε, να τρώνε προϊόντα τα οποία έχουν ε, πολλές θερμίδες, πολύ αλάτι ή πολύ λίπος. Δικό τους θέμα είναι. Απλώς πρέπει να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία στη διάθεσή τους για να κάνουν τις επιλογές τους. Όπως παραδείγματος χάρη όταν αγοράζει κάποιος αυτοκίνητο ή μια ηλεκτρική συσκευή του λέμε τι καταναλώνει όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια ή πόση βενζίνη χρειάζεται. Το ίδιο ισχύει και για τα, τρόφιμα. Οι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν τι αγοράζουν και θέλουν να τους αντιμετωπίζουμε με έναν έντιμο και δίκαιο τρόπο. Και τα, τα τρόφιμα είναι ένα προϊόν όπως όλα τα άλλα. Παραδείγματος χάρη για το κρασί θέλουμε να ξέρουμε ποιος είναι ο αλκοολομετικός τίτλος ε, του κρασιού και πόσες θερμίδες έχει ένα ποτήρι κρασί και πόσες θερμίδες έχει ένα ποτήρι ουίσκι ας πούμε ή κάποιο άλλο αλκοόλ, αλκοολούχο ποτό. Θα πρέπει δηλαδή οι επιχειρήσεις, οι τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να βρουν να επηρεάσουν τις τοπικές τους αγορές με αυτού του είδους τις πληροφορίες. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλά επίσης προϊόντα απομίμησης ε, και τα, για τα οποία πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα, όσον αφορά το κρέας, υπάρχει, υπάρχουν διάφοροι τύποι κρέατων που δεν έχουν τη σωστή σήμανση. Θα πρέπει τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση το κρέας να έχουν σωστή σήμανση. Ε, κάποια προϊόντα, για κάποια προϊόντα θα πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχονται. Π.χ. τα αυγά στα μεταποιημένα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ για τους συντηρητικούς. Κύριο Σίμωνσον, θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση κάποιων συστατικών. Παραδείγματο χάρη να είναι ένα κρέας, έχει παραχθεί με υψηλού επίπεδου προδιαγραφές, αν δεν έχει μεταφερθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα διάφορα συστατικά και τα διάφορα τρόφιμα επιλέγονται βάσει πολύ συγκεκριμένων διαδικασιών, στις οποίες βεβαίως συμπεριλάμβεται και η τιμή και ο τρόπος παραγωγής. Το κόστος λοιπόν είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το κόστος συσκευασίας. Το κόστος συσκευασίας το οποίο είναι ένα επιπλέον κόστος. Η επισήμανση λοιπόν η υποχρεωτική θα πρέπει να περάσει από μία συγκεκριμένη μελέτη συνεπειών και αντικτύπου, αξιολόγηση, έτσι ώστε να δούμε ποιο είναι αυτό το επιπλέον παραδείγματος χάρη κόστος. Η περιεκτικότητα για τα μεταποιημένα προϊόντα των διάφορων συστατικών. Για προϊόντα παραδείγματος χάρη όπως το ουίσκι, αυτό είναι καθοριστικό. Σήμερα υπάρχουν ουίσκι πολύ χαμηλής ποιότητας που έρχονται από την Κίνα ή από την ε, Ιαπωνία με ονόματα που θυμίζουν πολύ περισσότερο παραδοσιακές χώρες παραγωγής whisky της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες είναι παραπλανητικές. Και γι' αυτό και θα σας ζητήσω να στηρίξετε την τροπολογία 254. Ευχαριστώ πολύ. Για την αριστερά, η κυρία Λιωτάρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα θα πρέπει να διαλέξουμε στρατόπεδο την βιομηχανία των τροφίμων ή τον καταναλωτή. Εγώ θα υποστηρίζω το και επίσης θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα επιλέξουμε το χρωματικό κώδικα ή αν θα εμπιστευτούμε τη βιομηχανία. Θέλουμε μια ετικέτα που να επιτρέψει τον καταναλωτή να επιλέγει εν επιγνώση αν θέλει περισσότερο λίπος, λιγότερο λίπος, περισσότερο ζάχαρη, περισσότερη ζάχαρη, λιγότερη ζάχαρη κλπ. Γιατί όλο και περισσότερο οι καταναλωτές παραπλανούνται. Το 25% των πολιτών έχουν προβλήματα με την ανάγνωση των συσκευασιών. Αφού για τις ηλεκτρικές συσκευές ε, βρίσκουμε φυσιολογική την αναγραφή της ενεργειακής απόδοσης, δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην θεωρούμε το ίδιο φυσιολογικό να περιγράφεται η θρεπτική αξία και το θρεπτικό προφίλ. καλημέρα κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Ο κύριος Σκότα έχει τον λόγο για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, συνάδελφοι, καλούμεθα να ψηφίσουμε μία ε, έκθεση που αφορά την, πληροφορία των, ε, την πληροφόρηση των καταναλωτών. Ξέρουμε όμως ε, τι πληροφορίες θέλουν οι καταναλωτές. Η τελευταία δημοσκόπηση που έγινε από την Κομισιόν ίσως να μην είναι αντιπροσωπευτική για την προσοχή που δείχνουν οι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια για τα τρόφιμα τα οποία επιλέγουν. Η προέλευση αλλά και άλλα χαρακτηριστικά όμως γίνονται πάρα πολύ βασικά στοιχεία για την επιλογή του καταναλωτή. Γνωρίζουμε ότι οι επιλογές τις οποίες κάνουμε σήμερα θα επηρεάσουν τις αγορές του αύριο. Το ξέρουμε, το συνειδητοποιούμε αυτό. Οι καταναλωτές δεν πρέπει να καθορίσουμε ε, τι θέλουν οι καταναλωτές. Μήπως πρέπει να γίνει μια νέα δημοσκόπηση, μήπως θα πρέπει να έχουμε συνεχείς επαφές και συζητήσεις με τους καταναλωτές, να ξέρουμε τι θέλουν. Πρέπει να τους εκπροσωπήσουμε καλύτερα. Γι' αυτό είμαστε εδώ τώρα. Θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας την επιθυμία τους να εμπλακούν περισσότερο στην νομοθεσία. Μήπως θα πρέπει να δούμε τι, ε, μήπως κάποιες, ε, κάποιες πληροφορίες ε, που υπάρχουν στην, στις ετικέτες είναι είτε περιτές είτε παραπλανητικές είτε έχουν, αφορούν πληροφορίες που δεν θέλουν οι καταναλωτές που δεν επηρεάζουν τις επιλογές τους. δεν πρέπει να είμαστε πατερναλιστές αλλά να ακούμε τις ανάγκες τους. Ευχαριστώ κύριε Σκότα, ο κύριος Σέγγεντι έχει, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι για την ομάδα μου γενικώ ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η πληροφόρηση των καταναλωτών και οι πληροφορίες που αναφέρονται πάνω στην συσκευασία και πρέπει να είναι ο παραγωγό, ή ο μεταποιητής ε, ο οποίο είναι υπεύθυνο για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, για κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο. Επομένω, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να στηρίζεται στα χρώματα και που θα βοηθάει να ξεχωρίζουμε κατευθείαν τα πιο υγιεινά προϊόντα. Όμω, οι πολυεθνικέ, οι μεγάλε πολυεθνικέ, είναι οι υποχρεωτικές γιατί είναι, συγγνώμη, είναι υπεύθυνες για την διάδοση σε όλη την Ευρώπη, για την κυκλοφορία σε όλα την Ευρώπη προϊόντων κακής ποιότητας. Υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, το Σόντ, το Κόρα και άλλα σούπερ μάρκετ έχουν πλημμυρίσει την αγορά με κακής ποιότητας προϊόντα. Γιατί χρειαζόμαστε κινέζικα προϊόντα ή κάποια άλλα προϊόντα τα οποία είναι βλαβερά. Ε, δεν θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους, την ε, βιολογική καλλιέργεια, τους τοπικούς παραγωγούς που προωθούν οι ε, προϊόντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Γιούσο για 1,5 λεπτό. Πρόκειται για ένα εξαιρετική σημασία κανονισμό για του κατανοητέ και για την τροφιμική βιομηχανία. Διότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε ισορροπία στι ετικέτε που να περιλαμβάνει όλα όσα είναι απαραίτητα, χωρί όμω να είναι τόσο εξαντλητική ώστε να δημιουργεί πρόβλημα. Ε, συγχαίρω την εισηγήτρια για τι προσπάθειέ τη και συμφωνώ μαζί τη ε, στι βασικέ ε, γραμμέ τη εισήγησή τη. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι διατροφικέ ε, Η Κομισιόν δεν σεβάστηκε τον ε, συμβιβασμό που, στην οποία είχαμε ε, ε, την δέσμευση που είχε αναλάβει ε, για να εφαρμόσει αυτά, αυτό το προφίλ και αυτές τις διατάξεις μέχρι ε, το Δεκέμβριο του 2009. Χρειαζόμαστε μια εναρμόνιση και πρέπει να αποφύγουμε τα εμπόδια στην πραγματική λειτουργία της ε, ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Ό,τι αφορά τη χώρα η σημερινή νομοθεσία προβλέπει αυτές τις πληροφορίες να αναγράφονται όταν αν δεν αναγραφούν μπορεί να οδηγηθεί ο καταναλωτής σε παραπλάνηση, σε λάθος. το να πάμε πιο μακριά θα δημιουργούσε σημαντικό οικονομικό άχθο στις επιχειρήσεις χωρίς ε, περισσότερο ωφέλη για τους Γιατί η χρήση τώρα των διαφόρων γλωσσών η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία που δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα μέχρι τώρα. Μην ξανανοίξουμε τη συζήτηση γιατί μπορεί αυτό να μας οδηγήσει σε ε, επικίνδυνους δρόμους. Ευχαριστώ. Thank you, dear colleague. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μέσερ Childers για 1,5 λεπτό. Κύρια Πρόεδρε, πάνω από το 60% των Ιρλανδών είναι υπέρβαρη, η παχύσαρκη. Και αυτό το φαινόμενο δυστυχώς ε, το παρατηρούμε σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν για μια συγκεκριμένη κατάσταση, μια κρίση που οδηγεί και σε άλλα φαινόμενα, σε άλλες ασθένειες όπως ε, διαβήτη και άλλες πολύ βλαβερές συνέπειες για την υγεία. Η επισήμανση λοιπόν των τροφίμων είναι ένα πολύ απλό, διαφανές και παγκόσμιο σύστημα για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από αυτά τα βλαβερά φαινόμενα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναγράφονται όχι μόνο οι ζάχαρη, οι θερμίδες αλλά και άλλες προστικές ουσίες. Θα πρέπει την ίδια ώρα να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την πώληση βλαβερών τροφίμων και ουσιών. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να αντισταθούν στις ε, πιέσεις και να δουν αυτή την επισήμανση σαν ένα κόκκινο φως, μια ένδειξη που δίνουμε στους καταναλωτές για την κατανάλωση τροφίμων. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Κορίν Λεπάς, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ε, εγώ θα επικεντρώσω την προσοχή μου στα θέματα των χρωματικών κωδικών. Ε, μου λένε ότι είναι περίπλοκο το θέμα. Είναι ψεύδε, ψέμα αυτό, μπορούμε να το απλουστεύσουμε. Και ούτως ή άλλως είναι μια σωστή πληροφόρηση. Ε, Από την άλλη πλευρά μας λένε ότι θεωρούμε τους καταναλωτές με τον τρόπο αυτό ε, σαν παιδιά. Και όμως όχι, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών θέλουν αυτό τον χρωματικό, την χρωματική κωδικοποίηση αν θέλετε. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Θέλουμε να προσπίσουμε την ε, δημόσια υγεία και τους καταναλωτές ή θέλουμε να ε, υποστηρίξουμε τους, ε, τις βιομηχανίες και το λόμπι των, των κατασκευαστών που τον οποίων ούτως ή άλλως τα αιτήματά τους είναι και βραχυπρόθεσμα. Εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε τους ε, καταναλωτές. Ε, οι καταναλωτές ζητούν ε, τέτοιου είδους πληροφορίες για να διασφαλιστεί η υγεία στην Ευρώπη, γιατί είναι ένας τρόπος για να καταπολεμήσουμε την παχυσαρκία και διάφορες άλλες ασθένειες. Επομένως, μην λυγίσουμε, ας ξέρουμε για ποιους λόγους είμαστε εδώ, για ποιους λόγους μας έχουν εκλέξει, για να υπερασπίσουμε τους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ η κυρία Άση για ένα λεπτό. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν είμαστε αυτό που τρώμε, τότε είμαστε όλο και περισσότερο ένα βιομηχανικό προϊόν. Όλο και περισσότερους υπέρβαρους, όλο και περισσότερους παχύσαρκους, βλέπουμε όλο και περισσότερα καρδιακά προβλήματα και άλλου είδους ασθένειες το μοντέλο του, των χρωμάτων του σηματοδότη είναι απόλυτα κατανοητό ακόμα και από ένα παιδί με μια ματιά και μόνο. Αν δεν το εγκρίνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε τουλάχιστον τα κράτη-μέλη να επιτρέπεται να το χρησιμοποιούν σε εθελοντική βάση. Επίσης, για τα φυτικά λύπη τρανς θα έπρεπε να υποχρεωτικά να αναγράφονται. είναι σαφές ότι ε, επιβαρύνουν την υγεία και η παρουσία του στα τρόφιμα θα έπρεπε να αναγράφεται στις ετικέτες έτσι ώστε κάποιοι που αγοράζουν τσίπς ε, με σοκολάτα ή οποιοδήποτε άλλο σνακ να γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νίκολσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω την έκθεση και συγχαίρω την εισηγήτρια. Ασχολείται εδώ και αρκετό χρόνο και πραγματικά είναι πολύ ικανή ως ε, εισηγήτρια παράλληλα ότι δεν έχει πολύ χρόνο σαν βουλευτής. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σαφείς όταν μιλάμε για την, ε, για την ετικετοθυσία και για τα χρώματα. Προφανώς ε, θα πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής από πού προέρχονται τα προϊόντα. Επίσης ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πώς παρασκευάστηκε το τρόφιμο αυτό, το προϊόν αυτό. Επομένως συμφωνώ με την εισηγήτρια. Επίσης ε, πιστεύω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα πάρα πολύ νωρί Είναι μια διαδικασία, είναι η πρώτη ανάγνωση. Θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά πολλές φορές και αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να προχωρήσουμε συνετά, προσεκτικά, αλλά στο σωστό δρόμο. Δεν θέλουμε να υπάρχει μια υπερβολική νομοθεσία στην Ευρώπη και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί υπάρχει ένας ε, κίνδυνος αυτός να ε, ε, νομοθετήσουμε υπερβολικά, να μην ξέρουμε τι γίνεται. Γι' αυτό θα πρέπει το χρόνο ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ανάγνωση να το να τον χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μια μελέτη συνεπειών, να ξέρουμε πού προχωρούμε και τι έχουμε πετύχει ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ κύριε Νίκολσον, η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι κανείς εδώ θα πει ότι οι καταναλωτές ε, δεν θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα τρόφιμά τους και δεν θέλουν να είναι και ασφαλή. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πληθώρα πληροφοριών. Πρέπει οι πληροφορίες να είναι κατανοητές γιατί αλλιώς ο καταναλωτής αν έχει πολλές πληροφορίες δεν μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή του στις σημαντικές, σε αυτές που έχουν αξία. Αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριο επιλογής για τις πληροφορίες που μπαίνουν σε μια ετικέτα. Όσον αφορά την χώρα προέλευση, είναι σημαντικό να ξέρει κάποιο από πού προέρχεται ένα τρόφιμο που θα καταναλώσει. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες σήμερα που παράγουν τρόφιμα με πολύ αυστηρούς κανόνες. Ξέρουμε όμως ότι το 60% των τροφίμων εισάγονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι υπάρχουν κανόνες παραγωγής στις χώρες αυτές που δεν είναι καθόλου συγκρίσιμη με αυτούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Βόρεια Ιρλανδία. Ο τομέας ε, της παραγωγής ε, τροφίμων είναι πάρα πολύ σημαντικός και δεν θα πρέπει εδώ να επιβαρύνουμε τον τομέα αυτό με επιπλέον γραφειοκρατικό άγδος. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Φρανσουάζ Γκροστέτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ θα επιμείνω σε δύο θέματα. Πρώτον, το θέμα της διατροφικής δήλωσης. Προτείνω την διαγραφή της, διότι ο μοναδικός στόχος είναι αν να αναγνωρίζετε αν ένα τρόφιμο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγείας ή όχι. Όμως δεν θέλουμε να παραπλανήσουμε τον καταναλωτή με τέτοιου είδους ισχυρισμούς ε, οι οποίοι ε, μπορεί να ε, ε, ήταν χρήσιμοι κατά τα άλλα για τρόφιμα με υψηλό ποσοστό λίπους κλπ. Για το, για το άρθρο 205 τώρα. Δεν θέλουμε να στιγματίσουμε συγκεκριμένες θρησκευτικέ ομάδες, γιατί μια τέτοια ετικέτα θα δημιουργούσε ε, δυσπιστία, αβάσιμη δυσπιστία όμως. Γιατί ακόμα και τα τρόφιμα τα οποία είναι, ε, έχουν ε, σφαγή σύμφωνα με τα λειτουργικά έθιμα μπορεί να είναι εξαιρετικά υγιεινά. Πολύ περισσότερο προέρχονται από εγκαταστάσεις που είναι πιστοποιημένες και θα, μια τέτοιου είδου ε, ετικέτα θα μπορούσε να υποσκάψει την ύπαρξή τους ε, και βέβαια όχι μόνο των σφαγίων αλλά και των ε, παραγωγών εκτινοτρόφων. Σε ό,τι διαφορά αφορά τον χρωματικό κώδικα δεν πιστεύω ότι είναι σωστή λύση γιατί θα στιγμάτιζε τα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τον κύριο Περέγιο Ροντρίγκες. χίλιες τροπολογίες έχουν υποβληθεί και αυτό σημαίνει ότι, είμαστε, ότι έχουμε όλοι πολύ καλή θέληση να συνεργαστούμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Δεν θα πρέπει να παραπλανήνουμε τον κατανοητή, αντίθετα να τον βοηθούμε να αποφασίσει. Θα πρέπει να προλάβουμε παραπλανητικές πληροφορίες. θα πρέπει να αναγράφουμε αυτά τα οποία επηρεάζουν την χολυστερίνη, τα λίπη, τα τρανς, τα ζάχαρα κλπ. Ναι, εντάξει, αλλά περισσότερες πληροφορίες ίσως ε, θα δημιουργούσαν παραπλάνηση και σύγχυση. Ε, χώρα καταγωγής, χώρα προέλευσης, ε, χώρα σφαγής, χώρα που μεγάλωσε ένα ζώο, όλα αυτά ίσως είναι περιτά. Θέλουμε, πρέπει να αποφασίσουμε να αναγράφονται αυτά τα οποία θα βοηθήσουν τον καταναλωτή. Όχι θα να του δημιουργούν σύγχυση. Συνεπώς, εμείς προτιμάμε τις προς προσλαμβανόμενες ποσότητες και όχι τον ε, σηματοδότη. Γιατί να του βάλουμε κόκκινο σε έναν τρόφιμο το οποίο αν το φάει μια φορά δεν του κάνει τίποτα. Απλά του δημιουργεί πρόβλημα να το τρώει σε μεγάλες ποσότητες. Για ποιο λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Το λόγο τον έχει ο κύριος Chris Davis για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Τι θα ήταν απλούστερο από το να βάλουμε, να υιοθετήσουμε κανόνε που να δίνουν πληροφορίε στους καταναλωτέ. Υπάρχουν όμω διαφορετικέ ερμηνείε, διαφορετικέ πρακτικέ και συγκρουόμενα συμφέροντα σε διάφορε χώρε που ε, περιπλέκουν την κατάσταση. Τώρα για την σηματοδότηση ε, υπάρχει κάτι τέτοιο για τα ε, ενοπνευματώδη προϊόντα παραδείγματο χάρη. Όμως η πείρα που έχουμε μέχρι τώρα δείχνει ότι υπάρχει σύγχυση και υπάρχουν και διάφοροι ισχυρισμοί για την υγεία, ας πούμε, παραδείγματο χάρη. Με βάση από αυτά που άκουσα, υπάρχουν 44.000 ε, αιτήσει ε, που υπέβαλαν κάποιε ε, βιομηχανίε για ισχυρισμού για την προστασία τη υγεία. Ο οργανισμός για την υπηρεσία για, την, για, τα, για τα τρόφιμα έχει πλημμυρίσει, έχει κατακλειστεί από τέτοιου είδου αιτήματα και δεν ξέρουμε πώ θα βγούμε από αυτόν τον κικαιώνα και θέλουμε κάποια βοήθεια στη συγκεκριμένη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο τον έχει η κυρία Έμα Μακ για ένα λεπτό. Η αρχή για την αναγραφή περισσότερων και καλύτερων πληροφοριών για τον καταναλωτή είναι η αρχή ε, του κειμένου της οδηγίας. Όμως ε, συζητάμε πάρα πολύ ώρα για το τι θα αναγράφεται σε ένα μικρό πακετάκι με τσίχλες το αν το κοτόπουλο είναι πραγματικά κρέας ή όχι. Το σύστημα τον, ε, του σηματοδότη ε, υπεραπλουστεύει την, ε, τις διατροφικές δηλώσεις ε, και κατά βάση μειώνει τις επιλογές του καταναλωτή ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί πλήτη τον τομέα των προσκευασμένων των ε, τροφίμων πρώτης ανάγκης. Δεν μπορούμε περίπλοκες διατροφικές συνθέσεις, περίπλοκες συνθέσεις ε, τροφίμων να τις υπεραπλωστεύσουμε σε, ένα, σε τρία χρώματα. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι κατανοητές δεν θέλουν να τις επιβάλλουμε εμείς θα αγοράσουν και τι όχι. Αλλεργιογόνους, ουσίες ναι να τις περιλάβουμε αλλά όχι σηματοδότες. Τον λόγο τον έχει ο κύριος Μπόγκουσαν Σόνικ για 1,5 λεπτό. για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς η σήμανση των τροφίμων είναι ύψης της, ύψης της σημασίας. Επί του παρόντος υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες σε στα διαφορετικά κράτη-μέλη για τους ε, διάφορους κοινωνικούς κανόνες. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Με ανησυχούν ιδιαίτερα οι υποχρεωτικές πληροφορίες που αφορούν τη χώρα προέλευσης για κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Πιστεύω ότι κάποια κράτη-μέλη υποχωρούν ε, στον προστατευτισμό και ε, δημιουργούν ε, εμπόδια στην ελεύθερη αγορά. Η χώρα προέλευσης θα πρέπει να αναγράφεται ενημερωτικά έτσι ώστε ο καταναλωτής να προστατεύεται και ταυτόχρονα να προστατεύονται και τα συμφέροντα του κατασκευαστή. Μία ισορροπημένη διατροφή και ένας τρόπος ζω, σωστός υγιεινός τρόπος ζωής ήταν θέματα τα οποία ακούστηκαν διά, ε, πολλές φορές στην συζήτηση. Ε, όντως η σήμανση είναι ένα σημαντικός τρόπος ε, ενημέρωσης ε, των, και πληροφόρηση των καταναλωτών. Όμως μπορεί να γίνουν και άλλες εκστρατείες ενημέρωσης. Είμαι αντίθετος στην, στον σηματοδότη αυτόν, στον χρωματικό σηματοδότη, διότι θεωρώ ότι μπορεί να επηρεάσει και αρνητικά ακόμα την διατροφή στο κάτω-κάτω οι άνθρωποι αυτό το οποίο πρέπει να είμαστε σίγουροι είναι ότι είναι υπεύθυνοι για την επιλογή που κάνουν. Ο Κάρενμπακ για ένα λεπτά. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καθήκον των πολιτικών αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να εγγυηθούμε την ποιότητα ζωής και διατροφής των Ευρωπαίων πολιτών. Η υγεία των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τρόφιμα που καταναλώνουν και γι' αυτό χρειάζονται πληροφορίες. Επιγόντως λοιπόν χρειαζόμαστε μια δεσμευτική, μια υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης, της χώρας αλλά και της περιοχής προέλευσης για όλα τα τρόφιμα που αγοράζει ο καταναλωτής. Το διατροφικό προφίλ των τροφίμων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να παραπλανούν και να, να δίνουμε ελλειπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες η περιεκτικότητα κάποιων ουσιών είναι καθοριστική για την υγεία των καταναλωτών. Χρειάζεται την ίδια ώρα και καλύτερη εκπαίδευση στο τομέα της διατροφής και αυτό είναι κάτι το πολύ πιο μακροχρόνιο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο για ένα λεπτό έχει ο κύριος Κλούτσκι. Δεν συζητούμε πάντοτε νομοθετικά κείμενα που είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τους καταναλωτές μας. Αυτό όμως είναι ένα τέτοιο κείμενο και ασφαλώς οι επιλογές των καταναλωτών επηρεάζονται από την ε, επισήμανση των συσκευασιών. Ένα σημαντικό στοιχείο που, ε, το οποίο συζητάμε είναι οι πληροφορίες για, την, ε, για, τον, για τη χώρα προέλευσης των μεταποιημένων τροφίμων. Νομίζω ότι το, ο κανόνας του ότι αυτό θα έπρεπε να αναφέρεται στο βασικό συστατικό είναι πολύ καλός. Επίσης θα έπρεπε να αναφέρεται και η διατροφική αξία των αλκοολούχων προϊόντων ε, και όχι μόνο η διατροφική του αξία αλλά και ε, τα συστατικά ενός αλκοόλου ποτού. Ε, κάποιος πρέπει να ξέρει, για παράδειγμα, αν η βότκα που πίνει ε, είναι από πατάτα, είναι από μπανάνα, είναι από οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάολο Μπορτολότσι για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται, όπως ξέρουμε, να ε, πει την άποψή του, το οριστική του άποψη όσον αφορά ε, την ενημέρωση και τις προφορίες προς τους καταναλωτές. Πρόκειται για μια ε, νομοθετική διαδρομή η οποία ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη και που κράτησε αρκετά και, και δεν μπορούμε να την συντομεύσουμε διότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε την κοινοτική νομοθεσία μέσω των ε, της ρύθμισης ε, των ε, πληροφοριών που απευθύνονται στους καταναλωτές, κυρίως όσον αφορά πληροφορίες για προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι βλαβερά στην υγεία τους. Πραγματικά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυρία Σόμερ, διότι προσπάθησε να συντονίσει και να συμφιλιώσει διάφορες απόψεις και να εναρμονίσει τα διάφορα συστήματα τα οποία επικρατούν στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ε, υπάρχουν ε, πολλές νομοθεσίες ε, διαφορετικές σε κάθε χώρα όσον αφορά την ενημέρωση και τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στους ε, καταναλωτές. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια νέα πνοή, να, δώσει, να προτείνει νέα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και ενημέρωση των καταναλωτών. Επομένως, θα πρέπει και η, η βιομηχανία, η ευρωπαϊκή βιομηχανία να έχει σαφείς οδηγίες έτσι ώστε να δίνει και αυτή με τη σειρά της σαφείς οδηγίες και πληροφορίες προς τους καταναλωτές. Ε, και προφανώς Θα πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα και την ε, εμπορία των τροφίμων ε, στην, ε, που παράγονται στην Ευρώπη και να, να προστατεύσουμε τα προϊόντα αυτά από, τα, από τον σκληρό ανταγωνισμό που δέχονται από, από την διεθνή αγορά. Αυτό που προέχει είναι να έχουμε προϊόντα τα οποία να, είναι, να, να, να προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία. Ο κύριος Φερνάντες ε, για μισή λεπτό. Η επισήμανση των τροφίμων είναι ζωτική σημασία για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των τροφίμων. Οι πληροφορίε θα πρέπει να είναι σαφεί προ τον καταναλωτή, αλλά ταυτόχρονα να πρέπει να μειώσουμε και τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσουμε την νομοθεσία, να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και να μην ξεχνάμε ποτέ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η άμεση εμπορία από τους γεωργούς τοπικών προϊόντων δεν θα πρέπει να υπόκειται στο παιδί, να βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Γιατί αυτά τα προϊόντα έχουν σχέση με τις ρίζες μας, πιο βαθιές μας ρίζες. Θα πρέπει να ενημερώνουμε τον καταναλωτή χωρίς όμως να τον πιέζουμε στις επιλογές του ούτε να στιγματίζουμε τοπικά και ε, προϊόντα. Δεν θα πρέπει να είμαστε πατερναλιστικοί όπως το κείμενο, διότι ε, μάλλον όπως η πρόταση για τον σηματοδότη. Ποιος θα μας πει εμάς, θα ποιος θα μας επιβάλλει τι θα τρώμε και τι δεν θα τρώμε. εμείς δεν θα πάψουμε να τρώμε τα τοπικά μας προϊόντα, δεν θα πάψουμε να τρώμε τα δικά μας γιουβέτσια και τους δικούς μας μουσακάδες, επειδή κάποιος θα μας βάλει ένα φωτεινό σηματοδότη στο πακέτο. Συνεπώς, η συγγήτρια έχει δίκιο, ο καταναλωτής θα πρέπει να αποκτήσει συνείδηση να ενημερωθεί, να ενημερώνεται, αλλά ο ίδιος θα έχει την ευθύνη των επιλογών του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Φερνάντες. Τον, ρόλο, τον, τον λόγο του συγγνώμη τον έχει ε, η κυρία Μαγκίνες για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε για την ε, ενημέρωση για τα τρόφιμα. Ε, προς, ενημέρωση για τους, προς Το πρόβλημα δεν είναι, είναι τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες. Ε, καταρχάς ε, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως ας πούμε για το βόλιο κρέας υπάρχει κανόνας ε, που επιβάλλει την αναφορά της χώρας προέλευσης και που λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και όσον αφορά τα προϊόντα κρέατος, πιστεύω ότι χρειάζεται μια ανάγκη να υπάρχει πληροφόρηση για τη χώρα προέλευσης, έτσι ώστε να ξέρουν οι καταναλωτές από πού έρχεται το φαγητό τους. Απ' την άλλη πλευρά τώρα ε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, στο οποίο θα ήθελα να ρίξουμε φως. Ε, ευχαριστώ όλους όσοι μου έδωσαν πληροφορίες για αυτή την σηματοδότηση για το GDAs και προσπάθησα να αναλύσω τις πληροφορίες αυτές πάρα πολύ προσεκτικά και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, καταρχάς για τα στα τσιγάρα έχουμε προειδοποίησει όσον αφορά την υγεία. Εγώ δεν καπνίζω και πιστεύω ότι οι προειδοποίησεις είναι πάρα πολύ καλές αλλά εγώ δεν θα καπνίσω. Αυτοί όμως οι οποίοι είναι καπνιστές παρά τις προειδοποίησεις πάνω στα πακέτα συνεχίζουν να καπνίζουν. Επομένως δεν πρόκειται ούτε να σε βάλουν να σκεφτεί είσαι, ούτε, να σε, ούτε θα σε κάνουν να δυνατήσεις, ούτε θα, θα, θα πάψουν να σε κάνουν να είσαι παχύσαρκος. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι προφορίες που δίνουμε. Τώρα, στην πρώτη ανάγνωση έχουμε δει ότι ε, είναι, τα θέματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε τόσο γρήγορα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να ε, συζητήσουμε ε, με περισσότερες λεπτομέρειες όλες αυτές τις πληροφορίες που απευθύνουν τους καταναλωτέ. Ευχαριστώ. Τον λόγο τον έχει ο κύριος Ντόρφμαν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Πιστεύω ότι η επισήμανση των ειδών διατροφής είναι κάτι που αφορά όλους μας. Είναι κάτι που σαφώς και θα επηρεάσει τους καταναλωτές που ψωνίζουν είτε σε σούπερ μάρκετ είτε σε κάποια άλλα καταστήματα. Αυτό που όμως θα πρέπει να προσέξουμε είναι οι πληροφορίες αυτές να μην αλληλοεξοδετερώνονται και να είναι ουσιαστικές και να μπορεί να τις καταλάβει ο καταναλωτής. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι τα προϊόντα που είτε πολλούνται κατευθείαν από τους γεωργούς είτε πολλούνται και είναι προϊόντα παραδοσιακά χωρίς καμία απολύτως βιομηχανική ή άλλου είδους επεξεργασία. Παραδείγματος χάρη μαρμελάδες, ε, ε, γλυκά τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε αυτή την κατηγορία της ε, επισήμανσης και των υποχρεώσεων. Τα προϊόντα που πουλούν κατευθείαν οι γεωργοί στους καταναλωτές σε τοπικές αγορές είναι πολύ σημαντικό να προστατευτούν. Η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι κάτι που μας ε, απασχολεί σε άλλα πλαίσια και δεν θα πρέπει να τα ξεχάσουμε όταν μιλάμε για αυτήν εδώ την οδηγία. Η οι καταναλωτές που αγοράζουν κατευθείαν από τους γεωργούς θα πρέπει να προστατευτούν επίσης. Και αυτό είναι πιο σημαντικό από τις υπεχρεώσεις που επιβάλλουμε εδώ για την επισήμανση των τροφίμων. Παρακαλώ πολύ λοιπόν όλους τους συναδέλφους να προσέξουν και την πτυχή αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντόρφμαν, ο κύριος Ρίτσαρτ Ζέμπερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν θέματα υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και σαφώ και ο ρόλος του καταναλωτή όταν αγοράζει τρόφιμα θα πρέπει να ενισχυθεί. Τα προϊόντα αυτά δεν είναι ε, κοινά προϊόντα που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο άλλα προϊόντα. Έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία. Χρειάζεται λοιπόν εδώ μια διαφορετική ενημέρωση. Όταν μιλάμε για την επισήμανση των τροφίμων, βεβαίως δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Κοιτάξτε παραδείγματο χάρη τι γίνεται στην Αμερική, όπου η επισήμανση των τροφίμων είναι η πιο αυστηρή και η πιο λεπτομερής που υπάρχει στον κόσμο. Δεν έχουν προβλήματα υγείας και παχυσαρκίας στην Αμερική. Βλέπετε λοιπόν ότι η πληροφορία είναι σημαντική, η εκπαίδευση είναι ακόμα σημαντικότερη. Θα πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε τις πληροφορίες αυτές έτσι ώστε ο καταναλωτής να πάρει τη σωστή απόφαση. Και οι πληροφορίες στην ετικέτα δεν αρκούν γι' αυτό. Οι περισσότεροι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχεται το προϊόν που αγοράζουν και πού μεταποιήθηκε και πώς μεταποιήθηκε. Αυτό λοιπόν με έναν τρόπο κατανοητό. Επίσης, ο καταναλωτής θέλει να τον βοηθάμε να παίρνει την απόφασή του, να συγκρίνει δηλαδή μεταξύ συγκρίσιμων πληροφοριών, αλλά δεν μπορούμε να τον επηρεάσουμε. Επίσης ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές όσον αφορά τα στοιχεία αυτά και αυτές δεν θα πρέπει επουδενή λόγο να τις παρεκκλίνουμε και να τις αγνοήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σίμπερ. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε λάβει πολλές αιτήσει και βεβαίως δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε το λόγο σε όλους τους ομιλητές. Υπάρχουν πάνω από 15 αιτήσει μέχρι τώρα. Θα δώσω όμως αμέσως το λόγο στον ε, κύριο Βέσκερμπερ Άνια την κυρία Βέσκερ Μπερνάνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με αυτήν τη νέα πρόταση έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο μιας προσπάθειας να παρέχουμε στον καταναλωτή ενιαία στοιχεία, συγκρίσιμα στοιχεία, για να τον βοηθήσουμε να κάνει την επιλογή του θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα αποφύγουμε σφαλμένες και παραπλανητικές πληροφορίες για προϊόντα που είναι παραδείγματος χάριν ε, απομιμήσεις προϊόντων ή προϊόντα που είναι υποκατάστατα. Ένα γιαούρτι με γεύση βανίλιας που δεν περιέχει ίχνος πραγματικής βανίλιας. Όλα αυτά λοιπόν σαφώς και θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε να παρέχουμε νέα στοιχεία. Και όλοι συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε καλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή και όχι μόνο για τα τρόφιμα, αλλά τα τρόφιμα, όπως ξέρετε, επηρεάζουν άμεσα την υγεία. Είμαι λοιπόν υπέρ της καλύτερης επισήμανσης και πιστεύω ότι το σύστημα που προτείνεται αυτό εδώ είναι το καλύτερο και αύριο θα ψηφίσω υπέρ. Αν συμμετάσχετε θα πρέπει να περιορίσετε στο ένα λεπτό γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε. <laughs> Μιλάμε για σηματοδότηση. Εγώ θα είμαι το κόκκινο φανάρι και θα σας διακόπτω στο ένα λεπτό. Ο κ. Σταμπάτζη. Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουμε το πρότυπο που έχει υποβληθεί εδώ με τους σηματοδότες. Θεωρούμε ότι αυτό το μοντέλο, αυτό το πρότυπο θα μπορέσει να αποφύγει εσφαλμένες και λανθασμένες πληροφορίες και θα είναι προς του καταναλωτή. Με τα παραδοσιακά προϊόντα βεβαίως θεωρούμε ότι η σήμανση θα πρέπει να απευθύνεται μόνο σε κάποιες ειδικέ κατηγορίες προϊόντων. Όσον αφορά τη χώρα προέλευσης, θα πρέπει να υπάρχει κάποια πληροφόρηση, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει σε με τα ποιημένα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δίνω το λόγο στον κύριο Λαβία για ένα λεπτό. Εάν ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ε, ε, υγιεινά προϊόντα προς τους ε, καταναλωτές με έγκυρες πληροφορίες, αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση συστήματα σωστά επισήμανσης. Θα πρέπει να έχουμε ετικέτες που να έχουν πληροφορίες σαφείς και να ξέρει ο καταναλωτής ότι αγοράζει υγιεινή, προϊόντα, υγιεινά προϊόντα με έγκυρη προέλευση. Θα πρέπει να ε, επιστήσω την προσοχή σας σε ε, μια τροπολογία την οποία προσυπογράφουν 40 ε, βουλευτές, την τροπολογία 351, διότι θεωρούμε ότι θέλουμε, πρέπει να δώσουμε οπωσδήποτε στους καταναλωτές την προέλευση για την πρώτη ύλη και αυτό θα πρέπει να αφορά όχι μόνο κάποια γεωργικά προϊόντα αλλά και που, που έρχονται ως έχουν στην, από τις τρίτες χώρες αλλά και για τα ποιημένα προϊόντα. Ευχαριστώ. Τον λόγο τον έχει ο κύριος Ρίτς. Η κυρία Ρίτς. Ναι, η κυρία, κυρία Ρίτς, είστε εγγεγραμμένοι. Να μας δώσετε, να μας δώσετε τον κατάλογο των ομιλητών, όπως και για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, Υπάρχει ο κατάλογος όλων των, ε, των ομιλητών. Κυρία από την Άλντε, κυρία Ρίτσα. Ρώση, Μίστερ Πάσκα. Λοιπόν, αυτά τα ονόματα είναι τα αιτήματα τα οποία έχω, τα άτομα τα, άτομα οποία ζήτησαν να μιλήσουν. Λοιπόν, κυρία Ρίτσε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο πράγματα για αυτόν τον κανονισμό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιβεβαιώσουμε αύριο την υποχρεωτική αναγραφή της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων, όπως ισχύει για πάρα πολλά προϊόντα, για το ψάρι, για το, για, για το βόλιο κρέας ε, κυρίως μετά την, ε, ε, τις τρελές αγελάδες, γιατί πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό προωθούμε και βοηθάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εισάγουν κάποιες καινοτόμες διαδικασίες και πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις, τις διαδικασίες που βοηθούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι αυτές που περιπλέκουν τα πράγματα και επιβαρύνουν την κατάσταση ε, εδώ πρότεινε και η κυρία Γκροστέτ ε, κάτι που αφορά την, ε, τον παραδοσιακό τρόπο σφαγής. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό τιμωρούμε, αν θέλετε, τα, τα προϊόντα αυτά. Για, μιλάμε για τις σφαγές που γίνονται για θρησκευτικού λόγους. κυρία Ρόσετς. Πρέγω den europæiske forbruger er θα είμαι και εγώ καταναλώτρια και θέλω να ξέρω τι βάζω στο στόμα μου. Στη δική μου χώρα ξέρω από πού προέρχεται το κρέας, οι σαλάτες που καταναλώνω κλπ. Και οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τη σύνθεση των προϊόντων που τρώνε. Χωρίς να χρειάζεται να είναι χημικοί ή να έχουν πάρει μαθήματα διατροφολογίας. Το τι περιλαμβάνουν τα 100 μιλιλίτρα ή 100 γραμμάρια πρέπει να φαίνεται καθαρά στην εμπρόστια όψη. Δεν θα πρέπει να παραπλανήσουμε τον καταναλωτή με υπερβολικά πολλές πληροφορίες στην ε, ε, συσκευασία, αλλά ούτε και να επιβάλλουμε πολύ λεπτομερή αναγραφή στοιχείων σε μη συσκευασισμένα προϊόντα, ιδιαίτερα τα παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα. Πρέπει να προσέξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί θα χάσουμε πάρα πολλές τέσσερα εργασίας. Ευχαριστώ. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Η δύναμη του καταναλωτή είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Βάση έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών που αναγράφονται με σαφή τρόπο και χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε τον καταναλωτή στις επιλογές του. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας το διαφορετικό τρόπο ζωής, τις παραδόσεις και να βρούμε λύσεις πρακτικές, παραδείγματος χάρη για το θέμα του νοπού κρέατος. Υπάρχουν βεβαίως πολλές ε, εναλλακτικές ε, λύσεις, είτε να είμαστε πολύ αυστηροί στην πολιτική μας, είτε να επιλέξουμε την ελεύθερη επιλογή του καταναλωτή βάσει μιας ε, πληροφόρησης αξιόπιστης. Και αυτό είναι η επιλογή την οποία στηρίζω. Πρέπει να βασιζόμαστε στις πληροφορίες που έχουμε από τους επιστήμονες, αλλά να είμαστε και ευέλικτοι. Και θα πρέπει η αγορά να δείξει ότι γνωρίζουμε σήμερα και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για τα προβλήματα που δημιουργούν τα τρόφιμα στην υγεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρσένης έχει το λόγο. Και εγώ υποστηρίζω τη χρωματική σήμανση και θέλω να επισημάνω για ένα άλλο θέμα. Κάθε ώρα που περνά, 300 γήπεδα ποδοσφαίρου, έκταση ίση με 300 γήπεδα ποδοσφαίρου δασών, τροπικών παρθένων δασών, μετατρέπονται σε φυτίες φίνικα. Αυτό γίνεται προκειμένου να πάρουμε το φινικέλαιο το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή των τροφίμων που βρίσκουμε στα ράφια μας. Αυτή όμως η πληροφορία αποκρύπτεται από τους συμπολίτε μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλώ να υπεψηφίσετε την τροπολογία 263 που ακριβώς ε, αναφέρει ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ύπαρξης φινικέλου στα τρόφιμα που βρίσκουν οι συμπολίτες μας στα ράφια, ώστε να μην χρηματοδοτούν οι συμπολίτες μας την ε, παγκόσμια αποδάσωση την, την απώλεια της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το γνωρίζουν. Με την ψήφο μας αύριο, σε αυτή την αίθουσα, θα αποφασίσουμε αν οι πολίτες μπορούν να αναλαμβάνουν την περιβαλλοντική ευθύνη των διατροφικών τους επιλογών ή αν χρηματοδοτούν χωρίς να το θέλουν εταιρείες για να καταστρέφουν το περιβάλλον και το κοινό μας μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Όμπερμαϊερ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, οι μαθητές στην Ευρώπη σήμερα γνωρίζουν προβλήματα παχυσαρκίας σε πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε αυτό το θέμα και να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Είμαστε αυτό που τρώμε, αυτό που καταναλώνουμε. Η επισήμανση λοιπόν των τροφίμων είναι κάτι το πάρα πολύ ουσιαστικό. Είμαι λοιπόν υπέρ της ιδέας ότι θα πρέπει ο καταναλωτής με μια ματιά να βλέπει στην ετικέτα ενός προϊόντος που αγοράζει την περιεκτικότητα σε ζάχαρη, σε αλάτι και σε λιπαρά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει και την προέλευση των προϊόντων που αγοράζει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ενημερώνουμε τον καταναλωτή με τον τρόπο αυτό για το πόση απόσταση έχει διανύσει ένα προϊόν μέχρι να φτάσει σε αυτόν. Πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες οι οποίες είναι καθοριστικές. Υπάρχουν σήμερα συνέπειες. Αν δίνουμε εσφαλμένες πληροφορίες σε έναν καταναλωτή όσον αφορά την πρώτη ύλη παραδείγματος ενός μεταποιημένου προϊόντος, αυτό έχει άμεσες και σοβαρότητες συνέπειες στην υγεία του. Ευχαριστώ. Κυρία Κρίστα Κλάς. Σήμερα μιλάμε για πληροφορία, για ενημέρωση, κάτι το οποίο σήμερα δεν δίνεται απλώς με ελλειπή τρόπο, αλλά και πολλές φορές οδηγεί σε εσφαλμένες επιλογές. Σήμερα θα πρέπει να δούμε και το κόστος αυτής της σωστής και επιπλέον πληροφορίας. Η προσπάθεια για καλή ενημέρωση πρέπει να ξεκινήσει στις οικογένειες, στα σχολεία, στο εκπαιδευτικό σύστημα και είναι κάτι που θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο από την ψήφιση αυτής της οδηγίας. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό που προτείνει η σημερινή πρόταση έχει ε, και πάρα πάρα πολλές άσκοπες και άχρηστες πληροφορίες. Όσον αφορά τον σηματοδότη με τα χρώματα, δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα τον καταναλωτή να κάνει σωστές επιλογές. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι ένα τυρί μπορεί να παράγεται από γάλα που προέρχεται από ζώα που έχουν μεγαλώσει στο Λουξεμβούργο, κατόπιν το γάλα έχει μεταφερθεί στο Βέλγιο και το τυρί έχει παραχθεί στην Γερμανία. Βλέπετε λοιπόν ότι η προέλευση είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθοριστεί. Και αυτό ισχύει και για άλλα προϊόντα. Θα ήθελα λοιπόν να στηρίξουμε εδώ τις προτάσεις ε, της εισηγήτριας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάρμπο. Onorevole Sarbo. Non è presente l'onorevole Sarbo. Δεν είναι παρούσα η κυρία Γκρατσιάνα Σάρμπο. Το 638. No. Ok. Andiamo avanti. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Edith Estrella. Η κυρία Edith Estrella έχει το λόγο. Presidente, uma boa rotulagem μια καλή επισήμανση των ε, τροφίμων είναι ζωτική σημασίας. Ε, η αναγραφή του τόπου προέλευσης, ε, όπως επίσης και η περιεκτικότητα σε λίπη, σε ζάχαρη και σε αλάτι είναι απαραίτητα. Οι πληροφορίε αυτέ θα πρέπει να είναι ευανάγνωστε, σαφεί, προκειμένου να είναι αποτελεσματικέ. Να περιλαμβάνουν μόνο το απολύτω απαραίτητο. Όμω, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα έπρεπε ή δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν ορισμένα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία αποτελούν έκφανση μιας, ε, της κουλτούρας μιας συγκεκριμένης ε, περιοχής. Σε ό,τι αφορά το, τους ίνους, πιστεύω θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν και καλύπτεται από το δικό του κανονισμό. Δεν περιλαμβάνει ούτε ζάχαρη, ούτε λίπη. Περιλαμβάνει αλκοόλ του οποίου επιρρεκτικότητα αναφέρεται έτσι κι αλλιώς ε, στην, ε, ε, ετικέτα. Απ' την άλλη μεριά, η, μια καινούργιο τύπου επισήμανση θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα σε ένα τομέα ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει πολλά. Ευχαριστώ. Ρώσιο, κύριε Ρώσιο, αυτό το λόγο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία συνάδελφοι. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να γράφουμε την ε, προέλευση ε, των προϊόντων που εμείς καταναλώνουμε, εμείς και η οικογένειά μας. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία επιλογής, αλλά έχει δικαίωμα να ξέρει τι αγοράζει, τι έχει μέσα το προϊόν που αγοράζει και από πού προέρχεται. Πρέπει να δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία στον καταναλωτή να κάνει τις επιλογές του. Με αυτόν τον τρόπο το πρώτο βήμα για μια υγιή και ισορροπημένη ισορροπημένη δίαιτα είναι να ε, έχει τις απαραίτητες πληροφορίες ε, για να κάνει τις επιλογές του. Ε, δεν θα πρέπει όμως θα πρέπει μάλλον να έχουμε σε μια επισήμανση στα στοιχεία που θα επιτρέψουν που επιτρέψουν στον καταναλωτή να έχει την, ε, τις απαραίτητες πληροφορίες για να, κάνει, την, να πάρει την απόφασή του και όχι απλώς να λένε καλό ή κακό προϊόν. Πιστεύουμε ότι μια σωστή και ε, διατροφή ε, εξασφαλίζει και μια καλή ζωή. Κύριε Ρώση, μην τρέχετε τόσο πολύ όταν μιλάτε. Μια σύσταση απευθύνω, γιατί αλλιώς θα έχουμε προβλήματα όλοι και οι διερμηνείς ε, επίσης. κύριος Νικολέσκου έχει το λόγο. Subiectul codului de culori pare să fie cel mai aprins aspect al dezbaterii de astăzi. Το θέμα του σηματοδότη φαίνεται να είναι το πιο έτσι, επίμαχο. Ε, είναι αλκιστική ιδέα, αλλά σίγουρα δεν είναι αποτελεσματική και ενδεχομένω θα είναι και επικίνδυνη αν εφαρμοστεί. Δεν νομίζω ότι προωθεί την σωστή πληροφόρηση του κατανοτή. Ε, ε, δεν είναι δυνατόν να δαιμονοποιούμε τα συστατικά, το α το β συστατικό. Ε, δεν υπάρχουν κακά συστατικά, εξαρτάται το πόσο πολύ καταναλώνουμε κάθε φορά το κάθε συστατικό. Δεν θα πρέπει να παραπλανούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τον καταναλωτή. Ε, επίσης, συμφωνώ με τα όσα είπε η για τα κρέατα τα οποία είναι προϊόν ε, τελετουργικής θρησκευτική σφαγής με τελετουργικούς παραδοσιακούς ε, τρόπους. Δεν θα πρέπει να στιγματίσουμε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Επίσης, υποστηρίζω την 251 του κυρίου Λαβία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην προσπάθεια της εισηγήτριας να βελτιώσει την πρόταση της Επιτροπής. Βεβαίως και εμείς εδώ θέλουμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην καλύτερη ε, επισήμανση. Δεν μπορούμε να έχουμε πληθώρα ακατανόητων ε, στοιχείων, επιστημονικών ε, πληροφοριών, τις οποίες δεν μπορεί να καταλάβει ο καταναλωτής και τις οποίες προκαλούν σύγχυση. Πρέπει πραγματικά να είναι με σαφή τρόπο οι πληροφορίες αντικειμενικές, να είναι ακριβείς και οι διανομής θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το τι αναγράφεται σε μια ετικέτα. Πολύ φοβάμαι ότι η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το μέγεθος και την ευκρίνεια αυτών των πληροφοριών δεν είναι ικανοποιητικές. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο καταναλωτής να μπορεί με μια ματιά να καταλάβει τι περιέχουν αυτές οι πληροφορίες. Η επιλογή του καταναλωτή δεν μπορεί να γίνεται μόνο βάση της τιμής ενός τροφίμου. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς τη χώρα προέλευσης ενός προϊόντος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρόκειται εδώ για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, προστασία των καταναλωτών. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι η ασφάλεια των τροφίμων έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Ένας καταναλωτής σήμερα είναι πάρα πολύ δύσπιστο στην Ευρώπη η επισήμανση των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρέωση για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, τα χρώματα, ο σήμαδοτοδότης. Είμαστε υπέρ. Αν όμως αυτά τα χρώματα ακολουθούνται με τις διατροφικές αξίες και τα ποσοστά όπως τα ζητούμε. Επίσης, για τα υνοπνευματόδη ποτά και το κρασί. Ζητούμε μια ειδική ρύθμιση. Και αυτό θα πρέπει να γίνει τα τρία επόμενα χρόνια και όχι τα πέντε όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Νικολάσικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τη Ρενάτε Ζόμερ, γιατί ήταν δύσκολο το έργο της. Πρόταση αυτή είναι ένα σημαντικό νομοθετικό κείμενο για την υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Πολλές ε, ασθένειες είναι αποτέλεσμα κακών διατροφικών συνθήκων. Χρειάζεται λοιπόν μια συστηματική προσέγγιση οι κανονωτές θα πρέπει να διαθέτουν σαφείς πληροφορίες αλλά θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι τις επιλογές που τους αφορούν. Η δική μας δουλειά είναι να τους λέμε τι τρώνε και όχι τι πρέπει να τρώνε. Συνεπώς ε, το σύστημα του σηματοδότη είναι ανεπαρκές και επιδερμικό. 20% ε, των ε, επιχειρηματιών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν θα πρέπει να τους επιβαρύνουμε άλλο. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Επιτρόπο κύριο Ντάλι. Mr. President, honorable members. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήταν πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Η Κομισιόν θα μελετήσει προσεκτικά τις απόψει που ακούστηκαν. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους καταναλωτές κατά την άποψή μας. Πρώτον, η διαθεσιμότητα πληροφοριών για τα αλλεργιογόνα, ε, η ε, επισήμανση στην εμπρόστια όψη, μετρήσιμα κριτήρια για το επανάγνωστο και οι ισορροπημένες πληροφορίες ό,τι αφορά την υγεία υποστηρίζω την αρχή των ε, διατροφικών δηλώσεων και των ε, διατροφικών προφίλ και δεν θα σταματήσουμε την παραγωγή οποιασδήποτε, οποιοδήποτε μου. Θα είμαστε ανοιχτοί. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την διαγραφή της διάταξης αυτής. Θα ήθελα να απαντήσω όμως και σε ορισμένα σχόλια που έγιναν πιο συγκεκριμένα. Για την χρηματοδότηση θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε επί μιας μη νομοθετικής έκθεσης η οποία θα είναι έτοιμη μετά το καλοκαίρι και θα αναφέρει τις, τη γραμμή που θα ακολουθήσουμε. Σε ό,τι αφορά την καινοτομία, η προτάση μας δεν αντιδίκεται με την καινοτομία. Είμαστε υπέρ της καινοτομίας ασφαλώς ως Κομισιόν. Όμως θέλουμε την υπεύθυνη ευσυνείδητη καινοτομία υπέρ των καταναλωτών μας και υπέρ της υγείας των καταναλωτών μας. Σε ό,τι αφορά την οδηγία των ισχυρισμών, ε, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ντέιβις, υπό το άρθρο 30, ε, μάλλον το άρθρο, με βάση το άρθρο 30. Ε, λάβαμε 44.000 περίπου τέτοιες, τέτοιους Όταν ζητήσαμε τα κράτη-μέλη να τις εξετάσουν, ε, τις έκοψαν στις 4.000. Αυτό δείχνει ε, την, το ότι πολλές από αυτές, πολλοί από αυτούς τους χειρισμούς δεν ήταν σοβαροί, ήταν επιφανειακοί και ήταν απλώ ένα εργαλείο για να πολλούνται προϊόντα ε, προεργαλείο πρόθεση προϊόντων. Αυτό βέβαια καθυστέρησε τις διαδικασίες αρκετά, αλλά εργαζόμαστε επί της πρώτης ε, παρτίδα τέτοιων ισχυρισμών, ε, ετοιμαζόμαστε να την δημοσιεύσουμε και η δεύτερη θα ακολουθήσει. Δυνάμει του άρθρου 14 από την άλλη μεριά έχουμε 50 ισχυρισμούς, 50 ε, δηλώσεις ε, ε, οι οποίες έχουν ήδη κριθεί από την Κομισιόν. Συνεπώς και εκεί προχωράμε παρόλες τις καθυστερήσεις στο παρελθόν. Και θα ήθελα να κάνω άλλο ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά τις μελέτες ακτίμησης ε, ε, επιπτώσεων, αξιολόγηση επιπτώσεων. Εμείς ε, προέβημε σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και αξιολογήσαμε τον αντίκτυπο διαφόρων προτάσεων. Οι επιπτώσεις ορισμένων προτάσεων, στις οποίες αναφέρθηκαν ορισμένοι συνάδελφοι, δεν έχει δεν έχουν αξιολογηθεί. Πιστεύω ότι θα έπρεπε η διαδικασία εκτίμηση επιπτώσεων να ακολουθεί, να συνοδεύει την νομοθετική διαδικασία σε κάθε περίπτωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ζόμερ και του ε, βουλευτέ που έλαβαν το λόγο θέση της ε, Κομισιόν για κάθε μία από τις τροπολογίες είναι διαθέσιμη σε εσά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφου που πήραν τον λόγο και περνάμε στο, επόμενο σημείο η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων και αυξημένε ελεκτρικέ εξουσίες της Ευρώπης μέσω της Eurostat. Τον λόγο τον έχει ο κύριος Ότμαρ Κάρας για δυόμιση λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλοι ρε.